Dear colleagues, good morning. Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Εγκρίνονται την ημερήσια διάταξη της συνεδριάσεώς μας. Είναι μια ανοιχτή συνεδρίαση των συντονιστών. Είναι αφιερωμένη σε ανταλλαγή απόψεων με τον Κρίστιαν Τίμαν, τον καλωσορίζουμε. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε για δεύτερη φορά. Όπως ε, γνωρίζετε, θα μιλήσει στην Επιτροπή μας. Θα μας παρουσιάσει τις τελικές συστάσεις της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επίπεδου όσον αφορά το θέμα ενός βιωσίμου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Θα έχετε δει το κείμενο σε ηλεκτρονική μορφή, μια και θέλουμε να ακολουθήσουμε βιώσιμη προσέγγιση όσον αφορά τα ζητήματα των εγγράφων. Η έκθεση δεν περιορίζεται απλώς σε γενικές ε, πτυχές, αλλά υπησέρχεται εις βάθος θεμάτων. Δεν λέει μόνο τι πρέπει να κάνουμε και γιατί, αλλά και με ποιο τρόπο μπορούμε συγκεκριμένα το, την βιωσιμότητα, τη την πτυχή της βιωσιμότητας να την εντάξουμε στον χρηματοστατικό τομέα. Είναι πολύ καλή έκθεση. ετοιμάζουμε και τη δική μας έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας για το βιώσιμο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Ο Σκοσκέτερ είναι εδώ, θα πάρει το λόγο μετά την παρουσίαση, θα μιλήσουν και οι σκιώδεις και θα μπορέσουν οι συνάδελφοι να μιλήσουν και να υποβάλουν ερωτήσεις. Να δώσω το λόγο αμέσως στον Κρίστιαν Τίμαν που θα μας κάνει μια παρουσίαση. Θα διαρκέσει 10-15 λεπτά και μετά οι συνάδελφοι θα μπορέσουν να πάρουν το λόγο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Είναι μεγάλη χαρά για μένα που επιστρέφω εδώ. Ήμουν εδώ το Σεπτέμβριο και συζητούσαμε αυτά τα θέματα. Είχαμε μόνο ε, την ενδιάμεση έκθεση. Ήταν πολύ σημαντική αυτή η έκθεση ε, που δημοσιεύτηκε μόλις χθες. Πολύ σημαντικό η ομάδα μας. Ευχαριστώ για τις ανταλλαγές απόψεων που είχαμε. Μας ενέπνευσαν Προσπαθήσαμε πολλά από αυτά τα θέματα να τα λάβουμε υπόψη, διότι ξέρουμε ότι παρόμοιο ο προβληματισμό σα, παρόμοια η προσέγγιση σα, εξετάστε παρόμοια θέματα και θέλαμε να προσεγγίσουμε τι προσεγγίσει μα για να είμαστε όσο πιο δυνατόν ε, παραγωγικοί. Από ό,τι αφορά τιμή, όλα τα μέλη τη ομάδα υψηλού επίπεδου εργάστηκαν πολύ σκληρά. Ευχαριστώ του παρατηρητέ που με γενοδορία μα έδωσαν τον χρόνο του και την εμπρογνωμοσύνη του. Ήταν πολύ δραστήριοι. Ευχαριστούμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μα έδωσε εξαιρετική επιμελιακή υποστήριξη όσον αφορά τεχνικά ζητήματα. Θεωρήσαμε όλοι ότι ήταν μια υπέροχη εμπειρία η συνεργασία του τελευταίο δίμηνο. Αυτό που έχετε μπροστά σας είναι μια έκθεση, προσπαθεί να είναι το βασικό σχέδιο για, τα, για έναν βιώσιμο χρηματοστοτικό τομέα. Είναι μακροσκελής η έκθεση, διότι δεν υπάρχει μια και μοναδική λύση. Ένας διακόπτης και να περάσουμε και να έχουμε ένα σύστημα βιώσιμο από εκεί που δεν ήταν βιώσιμο, θα ήταν υπέροχο αν είχαμε τέτοιο διακόπτη, δεν έχουμε. Ε, ποια είναι η εξολογησή μα, ότι πρέπει να εξεταστεί όλη η, δημοσιο... πολιτική και οι κανονισμοί και να εντοπιστούν οι αναγκαίε αλλαγέ. Ποιο είναι το καλό, ότι δεν χρειάζεται να ξανακατασκευάσουμε το πλαίσιο, αλλά πρέπει να εξετάσουμε τι λεπτομέρειε και να δούμε αν υπάρχει κανένα πρόβλημα, κάποιο θέμα για τη βιωσιμότητα, αν κάτι πρέπει να αλλάξει. Γι' αυτό στην έκθεση βλέπετε βασικές συστάσεις που πιστεύουμε ότι έχουν προτεραιότητα. Μετά έχετε γενικές συστάσεις, εγκάρσεις, συζητήσεις ανά χρηματοστικό ε, τομέα, ε, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες κλπ. Και μετά ένα κεφάλαιο με γενικότερα θέματα, περιβάλλον, κοινωνία, ε, γεωργία, που πιστεύουμε ότι είναι σημαντικότατη τομή και ότι θα πρέπει αυτά τα θέματα να εξεταστούν. Οι δύο επιτακτικές ανάγκες για τον βιώσιμο χρηματοδοτικό τομέα περί πρόκειται. Δύο θέματα είναι βασικά. Το πρώτο, πρέπει να έχουμε ευρύτερη προσέγγιση, να ανοίξουμε τα μάτια μας και να λάβουμε υπόψη μας περιβαλλοντικές, κοινωνικές και κλιματολογικές πτυχές ευρύτερη προσέγγιση και προβληματισμό, να λάβουν υπόψη σχετικού κινδύνου και μετά μακροπρόθεσμη προσέγγιση και βιώσιμο χρηματοστικό τομέα. Τι σημαίνει ότι χρειάζεται φυσική επένδυση σε ανανόσιμε πηγέ ενέργεια, σε αλλαγέ στο σύστημα μεταφορών, αλλαγέ στον τομέα των αγροτροφημικών. τροφημικό, Άρα φυσικά αγαθά ε, που έχουν μια περίοδο απόσβεσης δεκαετιών θα πρέπει η χρηματοπιστωτική προσέγγιση να ευθυγραμμιστεί. Λοιπόν, ευρύτερη προσέγγιση και μακροπρόθεσμη ε, και οι σχετικές δράσεις. Θα δείτε τις βασικές συστάσεις. Οι βασικές συστάσεις, αν κατακλείδη, είναι καταρχάς να έχουμε μια ε, ταξονομία, δηλαδή να δούμε ποιοι τομείς είναι εκεί που απαιτούνται οι επενδύσεις. Αυτό για μας είναι η αφετηρία και θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τους επενδυτικούς ε, τομείς. Δεύτερον, χρειάζεται ξεκαθάρισμα όσον αφορά τα καθήκοντα τα επενδυτικά. Οι επενδυτές ε, πρέπει να εξετάσουν τους διάφορους κινδύνους και σε ποιο βαθμό και επί ποιας βάσος. Όπως ξέρετε, υπάρχουν διαφορετικά κύματα, διαφορετικές προσεγγίσεις όσον αφορά το θέμα και γι' αυτό προτείνουμε μία εναρμόνιση στην αντιμετώπιση των διαφόρων κινδύνων. Μετά χρειάζεται επίσης η αποκάλυψη στοιχείων να αναβαθμιστεί. Οπότε οι κίνδυνοι και ευκαιρίες που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα να γίνουν διαφανέστεροι όσον αφορά ε, την αποκάλυψη στοιχείων στους οικονομικούς φορείς. Τέταρτον, ε, προτείνουμε να δημιουργηθούν πρότυπα για την βιωσιμότητα ξεκινώντας με τα πράσινα ομόλογα. Αν υπάρχει ένα πρότυπο για τα πράσινα ομόλογα, αυτό θα προωθούσε όχι μόνο την αγορά, αλλά περισσότερες επενδύσεις στον τομέα αυτό. Και τελικά, όσον αφορά τι αστικέ θα ήθελα να τονίσω τις εποπτικέ αρχές. Πιστεύουμε ότι και αυτές θα πρέπει να εξετάσουν τα γενικότερα θέματα και να ενεργοποιηθούν ε, στις, και να τα λάβουν υπόψη στις συζητήσεις τους. Θα είδατε πολλές συζητήσεις που έγιναν. Εξετάσαμε κάποιες συστάσεις, θα αναφερθώ σε 7 σημεία, τα οποία θεωρώ ότι είναι πιο συγκεκριμένα και δεν είχαμε τη δυνατότητα να τα συζητήσουμε την περασμένη φορά και πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Καταρχάς, να, να δούμε την προσέγγιση τη βραχυπρόθεσμη. Υπάρχει ένα κεφάλαιο εκεί Γι' αυτό ε, το σκεφτήκαμε εκτενώς και οι συζητήσεις είναι ενδιαφέρουσες και οι απόψεις σας ε, θα ήταν πολυτιμότατες. Προσπαθήσαμε να κάνουμε, ε, εξετάσουμε τη βραχυπρόθεσμα χρηματοπιστωτικά στοιχεία με την προσέγγιση γενικότερη τη βραχυπρόθεσμη. Δεν είναι, δεν με τη διαχείριση της ρευστότητας και των αποθεμάτων και των ταμείων κλπ. Αλλά υπάρχει ένα θέμα όσον αφορά την βραχυπρόθεσμη προσέγγιση θεός των πραγμάτων. Προσπαθούμε να, το καθορίσουμε αυτό σαν να χρησιμοποιούμε μακροπρόθεσμα χρηματοδοτικά εργαλεία για να έχουμε βραχυπρόθεσμα ε, κέρδη. Μετοχές και ομόλογα είναι μακροπρόθεσμα ε, τέτοια ε, στοιχεία, αλλά προσπαθούν οι, αυτοί που τα χειρίζονται να έχουν βραχυπρόθεσμα κέρδη. Έχουμε όπως είναι το εμπόριο υψηλή συχνότητας. Όλοι αυτοί ε, κινούνται μέσα σε ένα μήνα, ότι είναι σε μια κλίμακα κάτω από ένα εξάμεινο και είναι πολύ δύσκολο και εκεί αυτό σχετίζεται με την οικονομική απόδοση. Προσπαθούμε να πούμε ότι χρειάζεται περισσότερη ανάλυση, να γίνει διάκριση μεταξύ βραχυπρόθεσμων προσέγγισης, άλλων πηγών χρηματοδότησης και να δούμε πού τα βραχυπρόθεσμα χρηματοπιστωτικά επηρεάζουν την πραγματική επένδυση και οδηγεί σε μείωση των επενδύσεων, διότι όλοι πιέζονται να δουν Πώ μπορούν να έχουν ε, βραχυπρόθεσμα κέρδη αντί μακροπρόθεσμε επενδύσεις. Και κάτι άλλο ε, εν είδη αγωγή. Είναι το θέμα τη βαθμονόμηση. Ξέρετε, οι χρηματοδοτικέ αγορέ καθορίζονται πολύ από αυτή την βαθμονόμηση για την παθητική επένδυση. Αλλά ε, βασιζόμαστε σε αυτή την βαθμολόγηση, την αξιολόγηση πάρα πολύ. Έχουμε τους διάφορους φορείς, Dow Jones, Φούτσι κλπ. Και η έκθεση τι αναφέρει, ότι πρέπει να έχουμε υπόψη ότι αυτό είναι υποσύνολο εταιριών και θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτό εδράζεται επί παρούσης αξιολογή της αγοράς. Αλλά ξέρουμε ότι η αγορά δεν λαμβάνει πλήρως υπόψη τους μελλοντικούς κινδύνους ε, και ευκαιρίες. Και αυτή η αξιολόγηση ίσως μην προσαρμόζεται με τον νέο κόσμο προς τον οποίο κινούμεθα. Οπότε ίσως να μην είναι οι σωστοί προσανατολισμοί και γι' αυτό έχουμε συστάσει στο σχέσμα να το εξετάσει αυτό το θέμα και να δει τι μπορεί να γίνει. Το τρίτο θέμα που θέλω να αναφέρω είναι τα λογιστικά. Εμπνευστήκαμε επίσης από τη δική σας συζήτηση και απόφαση ε, για το σχετικό κανονισμό και είπατε πιο συγκεκριμένο ότι θα θέλατε ε, να δείτε κατά πόσο ευθυγραμμίζονται τα μέτρα με μακροπρόθεσμες επενδύσεις ή όχι. Νομίζω ότι βρήκαμε επιχειρήματα στην έκθεση και ακούσαμε του εμπλεκομένου φορεί διάφορα που λένε ότι υπάρχει περιθώριο βελτιώσεων. βελτιώσεων. Το λέω και ελπίζω να χρησιμοποιώ τη σωστή διατύπωση. Το όλο πλαίσιο είναι καλό, αλλά υπάρχει ένα σημείο που είναι η αντιμετώπιση των διαφόρων αξιογράφων για μελλοντικέ επενδύσει. Αν οι μακροπρόθεσμε επενδύσει πρέπει να εκτίθενται ε, σε καθημερινές διακυμάνσεις ε, όσον αφορά το ισοζύγιο. Και έχουμε διάφορου τομείς που μας λένε ότι αυτό είναι αποθαρρυντικό για τη χρήση των αξιογράφων. Και αυτό επίσης επηρεάζει το, επηρεάζει το χρέος και την οικονομία. Κοιτάξτε, δεν μιλάμε κινητοποίηση ιδιωτικών πόρων, αλλά να βρούμε λογιστική προσέγγιση που θυγραμμίζεται περισσότερο με διάφορες ομάδες επενδυτών και έτσι θα ε, βελτιωθούν οι επενδύσεις. Τέταρτο θέμα, το τραπεζικό σύστημα συζητείται πολύ ο παράγων της υποστήριξης του πράσινου, πράσινης υποστήριξης, κάτι ευρύτερο. Έχουμε τον κανονισμό, τους κανονισμούς της Βασιλείας. Στη Βασιλεία συμφωνήθηκε ε, να καλυφτούν το που μας ενδιαφέρουν πολύ, διότι αφορούν τα το βιώσιμο χρηματοδοτικό σύστημα, ε, μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση, στεγαστικών δανείων, επενδύσεις μακροπρόθεσμες κλπ η συμφωνία της Βασιλείας συνήφθη ούτω ώστε να υπάρχει και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού παρόμοιο βάρος του κινδύνου. Αυτό ίσως αληθεύει, αλλά θα πρέπει να δούμε ότι οι Αμερικανικές τράπεζες δεν έχουν εισχωρήσει στο βαθμό που έχουμε εισχωρήσει εμείς στην Ευρώπη σε αυτόν τον κλάδο δεν είναι αρκετά σαφέ ότι μια διεθνή συμφωνία είναι καλύτερη, γιατί οι δραστηριότητε είναι φορετικέ. Οπότε η ομάδα συστήνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει προσεκτικότατα κατά πόσο αυτό πραγματικά είναι προ όφελο των ευρωπαϊκών μακροπρόθεσμων επενδύσεων, τη βιωσιμότητα και τη μακροπρόθεσμη δανειοδότηση. Το πέμπτο σημείο, και μετά έχω κανένα δύο, αφορά τον ασφαλιστικό τομέα. Υπάρχει ευρεία υποστήριξη όσον αφορά το Solvency 2 λειτουργεί πολύ καλά το πλαίσιο, όμως υπάρχουν ερωτηματικά για τα μακροπρόθεσμα προϊόντα και τη μακροπρόθεσμα αντιμετώπιση και έχουμε μακροπρόθεσμα πακέτο εγγυήσεων, πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει αυτό να επικυρωθεί. Δεν ξέρω αν μπορεί να κάνει κανείς περισσότερο για να τονώσει τις μακροπρόθεσμες, μακροχρόνιες επενδύσεις και μακροπρόθεσμα προϊόντα. Μετά είναι το θέμα των μετοχών, των λογιστικά ε, και επενδύσεις στα αξιόγραφα αυτό ωφελεί την, ε, τις παραγγελίες, μάλλον εκείνους που διαμορφώνουν την πολιτική και εκείνους που διαμορφώνουν τις επενδύσεις. Στο θέμα ε, της μετοχοποίησης θα πρέπει να το εξετάσουμε και να δούμε κατά πόσο μπορούμε να έχουμε ένα πλαίσιο κατάλληλο, πλαίσιο μετοχοποίησης διότι από, μπορέσουμε να μεταφέρουμε το τραπεζικό τομέα στον επενδυτικό. Μετά η οίκη αξιολόγηση. Θα δείτε ένα κεφάλαιο για τους οίκους αξιολόγησης. Δεν υπάρχει μεγάλη σαφήνεια σε ποιο βαθμό οι οίκοι αξιολόγηση λαμβάνουν υπόψη τη μακροπρόθεσμους κινδύνους και βιωσιμότητα στην αξιολόγηση. Μα λένε ότι την αξιολόγηση χρησιμοποιούν αυτοί που επενδύουν δύο-τρία χρόνια. Οπότε αυτά δεν είναι αρκετά σχετικά. Αλλά θα θέλαμε περισσότερο να τα εξετάσουμε αυτά και πιστεύουμε ότι η μακροπρόθεσμη περίοδο ξεκίνησε. εμεί είμαστε στη μακροπρόθεσμη περίοδο. Ακόμα μακροπρόθεσμα θέματα επίσης έχουν σημασία και σε βραχυπρόθεσμα ρίζοντα και θα τα εξετάσουμε αυτά και θα ενισχύσουμε και το ρόλο της, ε, ε, της βιωσιμότητας των οίκων αξιολόγησης. Και κάτι άλλο. Η ε, υποδομή ευρωπαϊκή, η καθεστική υποδομή στην Ευρώπη, Established Infrastructure Europe, βασισμένη στο σχέδιο Juncker, που ήταν επιτυχέστατο, κινητοποίησε επενδύσεις στον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά υπάρχει πολλή δουλειά να γίνει στον αφορά τις ε, υποδομές. Υπάρχει έλλειψη ε, ε δρομολόγηση των έργων. Οι ιδιωτικοί επενδυτέ όμω ε, περιμένουν. Δεν υπάρχει πρόβλημα ιδιωτικών επενδύσεων. Θέλουν να έχουν προϊόντα μακροπρόθεσμα υποδομών αλλά δεν υπάρχουν προγράμματα. Στην ανάλυση τι συμπεραίνει κανείς, ότι αυτό που λείπει είναι αναπτυξιακή δυναμικότητα. Αναπτυξιακή δυναμικότητα λείπει, ούτω ώστε τα κράτη-μέλη να αναπτύξουν διάφορα προγράμματα υποδομών. Εδώ μιλάμε για νέε τεχνολογίε, ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, αιωλική ενέργεια ε, ε, ε, και μεταμόρφωση του μεταφορικού τομέα και χρειάζεται δυναμικότητα. Εμπνευστήκαμε λοιπόν από τον Καναδά, όπου υπάρχει το Infrastructure Canada, μια υποδομή με 350 ανθρώπους που εργάζονται εκεί και αναπτύσσει διάφορα προϊόντα υποδομών σε όλη την Ήπειρο. Στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε την Infrastructure UK με 150 υπαλλήλους. Άρα, συγκεκριμένοι φορείς ή δίκτυα που πραγματικά βοηθούν τα κράτη-μέλη ούτως ώστε να αναπτύξουν διάφορα έργα υποδομών που προωθούν τη βιωσιμότητα στον οικονομία Αυτά λοιπόν ήθελα να τονίσω, απλώς εν είδη στη συζήτησή μας, θα σταματήσω εδώ και προσβλέπουμε στις απόψεις σας και σε προτάσεις σας. Ευχαριστώ για τα προηγούμενα σχολιάσατε, βίβασα στην ομάδα. Πολλά μέλη της ομάδας παρακολούθησαν, πολύ παρακολούθησαν τη συνεδρίασή μας και αυτό βοήθησε πολύ την ομάδα μας και ελπίζω να συνεργαστούμε, να συνεργαστείτε εσείς με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τους ώστε τελικά να προωθηθεί ένας βιώσιμος χρηματιστικός τομέας. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Θαυμάσια δουλειά έχετε κάνει και έχετε υιοθετήσει μια συνεπή προσέγγιση που από τη μία λοιπόν ε, έχει εσωτερική συνοχή αλλά και παρκές σημείο διαφορετικότητας που μας επιτρέπει να στοχεύσουμε με φιλόδοξο αλλά και ρεαλιστικό τρόπο τις λύσεις. Γιατί ξέρετε, μια μικροπροσαρμογή ε, σε ένα σημείο μπορεί να αλλάξει όλη την ισορροπία του μηχανισμού παροχής κινήτρων. Πολύ σωστή λοιπόν προσέγγιση και θα την εξετάσουμε και θα τη σχολιάσουμε. Πριν δώσω το λόγο στην εισηγήτρια, δύο παρατηρήσεις. Η πρώτη σχετίζεται με τη δουλειά που κάνουμε για τον τραπεζικό τομέα, όχι μόνο στον τομέα που εξετάζει η εισηγήτρια, που είναι μακροπρόθεσμη επενδυτική στρατηγική που μπορεί και πρέπει να σχετίζεται με την βιωσιμότητα. Τώρα που προετοιμάζουμε και την ψηφοφορία θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να αναπροσαρμόσουμε τον κανονισμό της Βασιλείας αν και η προσέγγισή μας είναι κάπως γενικότερη. Αλλά μπορούμε να αρχίσουμε να εργαζόμαστε και για κάποιους μηχανισμούς και στοιχεία στήριξης. Θέλαμε τη γνώμη σας γι' αυτό. Δεύτερον, πολύ πιστικός είναι αυτός ο πίνακας του κανονισμού για τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς και θα μπορούσαμε να το εξετάσουμε και να ζητήσουμε ε, από την Κομισιόν να κάνει κάτι γι' αυτό. Νομίζω ότι ενδιαφέρει την Pervance ε, Και η χρήση των αξιογράφων για... Αυτό εννοώ, η χρήση των αξιογράφων για μακροπρόθεσμες επενδύσεις στο πλαίσιο του IFRS. Θυμάστε επίσης ε, ότι την προηγούμενη φορά αναφέρθηκα και στην κοινωνική διάσταση της βιωσιμότητας. Δεν το αναφέρατε συγκεκριμένα, αλλά το έβδομο σημείο που αναφέρατε συνδυάζεται άψογα με την πρόσφατα δημοσιευθής έκθεση πρώτη για, την κοινωνική υποδο... για τις κοινωνικές υποδομές. Πώς θα βοηθήσουν τα διαφορετικά ταμεία και οι διάφορα άλλα στοιχεία, τα οποία με μικροπροσαρμογές θα μπορούσαν να βοηθήσουν πολύ την ανάπτυξη κοινωνικών υποδομών Όλα αυτά ενδιαφέρουν και στα πλαίσια της ε, βιωσιμότητας. Και πραγματικά είναι μακροπρόθεσμα. Τίποτα δεν είναι λιγότερο μακροπρόθεσμο από μια τέτοια προσέγγιση. Εδώ μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν ε, ενάρετο κύκλο μεταξύ των οικονομικών και κοινωνικών αναγκών αν υπάρξει ευφυής ε, συνδυασμός δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων κτλ. Τώρα, Κάτι άλλο. Ένα θέμα που αφορά τα δημοσιονομικά. Χρειάζεται ένα ε, σταθερό πλαίσιο που να ευνοεί τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Αυτό θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας όταν, και τους όταν αποφασίζουμε και τους φορολογικούς μας κανόνες. Εδώ χρειάζεται διαφοροποίηση. Προσπαθούμε να την εισαγάγουμε, αλλά δεν είναι ακόμη επαρκή να γίνεται σωστή διάκριση των επενδύσεων. Τι είδου επενδύσει είναι. Και να δίδονται τα κατάλληλα κίνητρα. Ξέρω ότι δεν σας αφορά άμεσα, αλλά εμείς εργαζόμεθα σε αυτούς τους τομείς και θα θέλαμε και από αυτόν τις απόψεις σας. Γιατί και αυτός ο τομέας θα πρέπει να διερευνηθεί. Ίσως στο τέλος θα μπορούσατε να σχολιάσετε. Αλλά πρώτα απ' όλα να δώσω το λόγο στην συγκήτριά μας, την Μόλι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς ε, να πω ότι είναι καταπληκτική έκθεση. Θαυμάσια δουλειά έχει κάνει η Επιτροπή σας. Νομίζω ότι είναι ιστορική σημασία. Και πραγματικά με συγκινεί να βλέπω κάτι τόσο σημαντικό για το μέλλον του πλανήτη και για τις μελλοντικέ γενιές και να βλέπω ότι ανταποκρίνονται στην πρόκληση αυτή τα μέλη της ομάδας σας. Παρακαλώ να τους μεταβιβάσετε τις ε, ευχαριστίες και τα συγχαρητήριά μου. Πρώτα απ' όλα κάτι το οποίο ίσως να ενοχλήσει. Γιατί δεν το είχα, δεν είχα όλα αυτά ε, ε, Αλλά ξέρετε ότι μια τόσο μεγάλη έκθεση είναι λίγο δύσκολη να μελετηθεί. Γιατί πρέπει να βασιζόμεθα σε αρχές, αλλά πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές. Ξέρουμε τις αρχές μας, αλλά πρέπει να δούμε και πώς θα τις εφαρμόσουμε συγκεκριμένα στις διάφορες φάσεις της μετάβασης στην βιωσιμότητα. Αυτό ισχύει για όλες τις εργασίες μας για τη βιωσιμότητα αλλά και για το βιώσιμο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Είναι λοιπόν μια διαδικασία μετάβασης. Δεν πρόκειται να καταλήξουμε απευθείας όλες τις σωστές λύσεις και να μείνουμε σε αυτές ε, ε, αδιάλακτα. Πρέπει λοιπόν να διευρύνουμε, μας λέτε, την έννοια της βιωσιμότητας, να μην βασίζεται μόνο σε κλιματικά κριτήρια. Και όταν συζητήσαμε το πώς θα αξιοποιήσουμε τα στοιχεία του ενεργητικού μας, το συνδυάσαμε με το κλίμα. Αλλά υπάρχουν χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι και σε άλλες διαστάσεις οικολογικής κρίσης. Για παράδειγμα, η εντατική γεωργία, επειδή συμμετέχω ε, και είμαι μία από τις λίγες και στην ΕΚΟΝ και στην Άγκρη, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Επίσης ε, μου αρέσουν πολύ οι προτάσεις σας για μία πολύ σωστή ιεράρχηση που να μπορούν να την καταλάβουν και οι επενδυτές για να μπορούμε ακριβώς να δίνουμε, να βαθμολογούμε όλα τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Θα πρέπει βέβαια να δούμε πώς θα λειτουργήσει όταν κατόπιν θα υπάρξει νομοθετική πρόταση από αυτού. Αλλά αυτή είναι η σωστή προσέγγιση, συμφωνώ. Και τέλος, Μ' αρέσει το κομμάτι σας για τις υποχρεώσεις των επενδυτών και καλύτερη πληροφόρηση προς τους επενδυτές μου είπε ότι εγώ δουλεύω σε μία ΜΚΟ για θέματα βιωσιμότητας και θα ήθελα να κάνω ε, βιώσιμες επενδύσεις, αλλά δεν ήξερε πώς να αξιοποιήσει την πληροφόρηση που έχει. Βεβαίως, θα πρέπει οι υποχρεώσει των επενδυτών να είναι σε όλη την αλυσίδα. Και τώρα να σας πω ορισμένα θέματα όπου έχω αμφιβολίες. Πρώτον, δεν θέλετε να είναι υποχρεωτική η γνωστοποίηση των κινδύνων για το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα. Το Κοινοβούλιο θα πιέσει γι' αυτό, είναι στην έκθεσή μα. Θέλουμε βεβαίω να δούμε πόσο θα το προχωρήσουμε μέσω των ε, διαπραγματεύσεων εντό του Κοινοβουλίου. Είπατε ότι πρέπει να αναβαθμιστούν οι περιπτώσει όπου θα γνωστοποιούνται οι κίνδυνοι. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει υποχρεωτική γνωστοποίηση αυτών των κινδύνων. Στα πλαίσια και τη μη χρηματοπιστωτική ε, υποχρέωση υποβολή εκθέσεων. Ήταν μεγάλη εκθεσή σα να μην τα διάβασα όλα. Αλλά νομίζω ότι ε, εστιάζεται Κυρίω στα δικά μα εσωτερικά όργανα χρηματοδότησης. Αλλά εγώ ανησυχώ για κάποιε από τι επενδύσει από την Τράπεζα Επενδύσεων που εξακολουθούν να είναι προς καύσιμα. Και θεωρούμε ότι το πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού και από τι εταιρείε αγοράζει τέτοια στοιχεία η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μας δημιουργεί ανησυχίε. Και κάτι άλλο που είναι πιο διαδικαστικό. Βεβαίω, είναι μακρόπνοη αυτή η προσπάθεια, το εγχείρημά σας. Αλλά Πώς θεωρείτε ότι παρόλα αυτά θα μπορούσαμε κάποια στοιχεία να μπουν στο θεσμικό πλαίσιο, ούτω ώστε όταν θα αλλάξουμε εμεί ως πολιτική και θα αλλάξει η Κομισιόν, να διατηρηθεί αυτή η κατεύθυνση. Πρόεδρος, εσύ παπιέτη τι κάναν. Ευχαριστώ. Για μία ακόμη φορά ευχαριστώ, κάνατε υπέροχη δουλειά. Ίσως μεροληπτό, αλλά ήταν η καλύτερη ομάδα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια δεκαετία. Κατεβλήθησαν πολλές προσπάθειες, ευφυής προβληματισμός και συγκεκριμένες εφαρμόσιμες προτάσεις έγιναν και κυρίως στο σωστό επίπεδο. Δεν θα αναφερθώ εκτενώς στις ιδέες όπως είναι η βαθμολόγηση και για την βραχυπρόθεσμη θεώρηση των πραγμάτων σημεία στα οποία πρέπει να εστιαστούν οι προσπάθειές μας. Έχω ελπίδες, επιθυμίες και ε, κάποια παράπονα όταν εξετάζω ένα κείμενο. Καμιά φορά όταν εστιάζεται κάποιος σε αυτά, λησμονεί ότι το μεγαλύτερο κομμάτι του κειμένου είναι καλό και κολλάει στα παράπονά του και στα δύσκολα σημεία αυτά που επιδέχονται βελτίωση. Δεν είναι πολλά σημεία που θα αναφέρω καινούρια για σας, ούτε την ομάδα εργασίας. Τα έχουμε συζητήσει και προηγουμένως. Αλλά θα ήθελα να περιγράψω τα σημεία που μας προβληματίζουν, διότι σε κάποια σημεία ίσως ε, άθελά μας να ακολουθούμε στραβόδρομο, ξεκινώντας από εκεί. Είναι η γενική συζήτηση για τους δείκτες. Κατανοώ ότι απαιτείται ποια, ποιος είναι, ποια είναι η πράσινη προσέγγιση και η πράσινη αξιολόγηση. Αυτό όμως είναι στο περιθώριο των συνολικών επενδύσεων που γίνονται στην Ευρώπη και παγκοσμίω. θα πρέπει να, να υπάρξει μια σωστή προσέγγιση όσον αφορά το πρασίνισμα της οικονομίας. Λοιπόν, η ανάπτυξη αυτής της ιεράρχησης συμπεριλαμβάνει την, τον προβληματισμό που ακολουθήσατε, αλλά θα ήθελα πιο ξεκάθαρα σημεία όσον αφορά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την προσέγγιση του Κοινοβουλίου ότι μας χρειάζονται κοινοί δείκτες ε, προς όπου θα λαμβάνει υπόψη την κατανάλωση πρώτων υλών, τις επιπτώσεις για το περιβάλλον και κοινωνικές επιπτώσεις. Και αυτές οι πτυχές να συμπεριληφθούν στο δημοσιονομικό κανονισμό, στην αξιολόγηση των επενδύσεων, βαθμολόγηση των επενδύσεων και στο IFRS να υπάρχουν συγκρίσιμε πληροφορίε για τον επενδυτή να ξέρει που είναι επενδύσει. Ποιο είναι ο φόβο μου? Ότι αν δεν ξεκινήσουμε σύντομα αυτή τη δουλειά και δεν έχουμε εργαλεία διαφοροποίησεως στον τομέα, τα διάφορα στοιχεία, είναι εύκολο να πει κανείς ότι μια επένδυση είναι καλή όσον αφορά την πράσινη προσέγγιση. Θα πρέπει να υπάρχει και διαφοροποίηση και των πετελαϊκών ε, εταιριών. Κάποιες κάνουν σωστές επενδύσεις για το πρασίνισμα της οικονομίας και κάποιες όχι. Και υπάρχουν κάποιοι δείκτες. Το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι εναρμονισμένοι. Αν δεν αρμονιστούν οι δείκτες. Αν δεν είναι υποχρεωτική εφαρμογή τους από όλους, δεν έχουμε συγκρίσιμα στοιχεία. Και δεν αλλάζει αρκετά γρήγορα το μεγαλύτερο ποσοστό των επενδύσεων. Δεν αλλάζει η ποσοστή κατεύθυνση. Τώρα, η υποχρεωτική αποκάλυψη στοιχείων. Γνωστοποίηση στοιχείων. Αυτό είναι κρίσιμη σημασία και θα, θα πρέπει να θεωρηθεί σαν ευθύνη, όπως η χρηματοδοτική ευθύνη θα πρέπει τα συστήματα να υπάρχουν σε μια επιχείρηση. Και θα πρέπει να υπάρχουν και έκθεσεις ελέγχου, να γίνεται ο έλεγχος. όσον αφορά τις επενδύσεις και τις πιστώσεις, τα στοιχεία ενεργετικού και άλλα συναφή στοιχεία. Ο δημοσιονομικός κανονισμός. Με αυτούς τους δείκτες θα έπρεπε να προβλέπετε ρήτρα αναθεώρησης. Όταν αναθεωρούνται οι δημοσιονομικοί κανονισμοί θα εξετάζονται κατά πόσο κάποιοι δείκτες είναι διαφανείς, λαμβάνουν υπόψη πράσινες πτυχές κλπ. Αυτό εν μέρει αναφέρεται στην έκθεση. Θα ήθελα όμως πιο σαφή διασύνδεση με τους δείκτες. Μετά επιδοτήσεις και οι στρεβλώσεις που μπορεί να προκαλέσουν στις χρηματοστατικές αγορές οι επιδοτήσεις και κυρίως όταν χρησιμοποιούμε ιδίους πόρους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και δημόσιες επενδύσεις και κρατικές προμήθειες. Θα πρέπει να ενταχθούν στον βιώσιμο χαρακτήρα. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούμε 20% του ΑΕΠ μας σε μη ε, βιώσιμες επενδύσεις. Ευχαριστώ για τους σοσιαλιστές. Υπερβάμος. Ο Πέτερ ζήτησε το λόγο, αλλά μπορεί στο Catch the Eye να λάβει το λόγο. Εκτός αν εγκαθιστά τον Πολ. Ποιος θα μιλήσει εκ μέρους του Πολ. Πρώτα υπερβάμος. Well, thank you very much. I mean, you've been doing great... Ευχαριστούμε πολύ. Έξοχη δουλειά σας. Σας βοήθησε όλη η εξέλιξη στον πλανήτη και η μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση, η βελτίωση της συνειδητοποίησης των προβλημάτων στον πλανήτη. Βλέπω να αλλάζει το πνεύμα και εδώ στο Κοινοβούλιο. Δεν το είδα ποτέ στο παρελθόν και σε κανένα άλλο τομέα. Δεν ενδιαφερόταν πολύ ο κόσμος αρχικά αυτή την ιδέα, ανακάλυψαν όμως τελικά ότι ενέπνευσε τελικά και τον τομέα των χρηματοπιστωτικών. Όμως πρέπει να γίνει δουλειά. Ευχαριστώ επίσης που λάβατε υπόψη την Βασιλεία. Κάθε φορά που συναντιόμασταν το ανέφερα αυτό και σας είπα αν δεν συμπεριλάβετε την Βασιλεία θα λείψει κάτι και τα ζητήματα που εξετάσατε όσον αφορά τα πρόσφατα αποτελέσματα της Βασιλείας δείξανε πόσο σημαντική είναι η ευρωπαϊκή φωνή που θα πρέπει να στηρίξει τα επιχειρήματά της περί βιώσιμου χρηματοπιστωτικού τομέα όταν διαπραγματεύεται. Όσον αφορά τον ασφαλιστικό τομέα, αναφερθήκατε στο Solvency 2, στη Φερικαιότητα 2. Το Solvency 2 ολοκληρώθηκε όταν οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις ποτέ δεν είχαν τεθεί επιτάπητος. Το προθούσαν αυτοί που δεν είχαν συναυθεί η συμφωνία, αλλά τελικά επευλήθη η δυναμική εκείνων που ήθελαν να διαπραγματευτούν επεκράτησε διαπραγματευτική κόπωση και ήθελα να ολοκληρωθούν διαπραγματεύσει. Αν θα ξανανοίξει η διαπραγμάτευση, πότε και πώ, δεν ξέρω. Θα γίνει μεγάλη αναθεώρηση στην επόμενη θητεία, αλλά α προετοιμαστούμε. Δεν θέλω τώρα να αναφερθώ σε όλα τα αναφερθέντα σημεία, είναι πολλά. Θα εστιαστώ επί δύο-τριών σημείων. Το πρώτο αφορά την βαθμολόγηση και την αξιολόγηση. Στην έκθεσή σας δεν εστιάζεσαι τόσο στις λεπτομέρειες της νομοθεσίας που εξετάζουμε. Αν θέλουμε να είμαστε επικοδομητικοί και ένας από τους λόγους που είμαστε εδώ είναι αυτός, είναι ότι εσείς τώρα εξετάζετε το πώς όλα αυτά μεταφράζονται σε νομοθεσία, όχι μόνο η ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα έχει ένα πλήρες πακέτο, θα μας δώσουν κάποια σημεία, θα αφήσει κάποια άλλα για την επόμενη θητεία, την εκστρατεία κλπ. την προεκλογική. Εν μεταξύ έχουμε πλήρες φάσμα ε, θεμάτων επιτάπητος που μπορεί να μας εμπνεύσουν ή και να εφαρμοστούν μέσω των στάσεων. Για τη βαθμολόγηση είναι το πρώτο παράδειγμα θα πάρω. Έχουμε στην αναθεώρηση ΕΣΑ, έχουμε έχουμε δημιουργήσει ένα πλαίσιο εκεί που θα πρέπει να ενταχθούν αυτά. Δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα όμω. Η βιωσιμότητα αυτή του χρηματοστικού τομέα δεν είναι κάτι εύκολο. Στα πλαίσια τη ΕΣΑ δεν θα κάτι, στην εντολή τη ΕΣΑ δεν θα είναι κάτι εύκολο. Μην το θεωρείτε δεδομένο λόγω τη εκθέσεω. σα. Βοηθήστε με να το στηρίξουμε αυτό. Δεύτερον. Και απογοητεύτηκα λίγο. Πρέπει να το ομολογήσω αυτό. Όσον αφορά την ιεράρχηση των θεμάτων επιμακρών συζητούμε εθελοντική υποχρεωτικά κριτήρια, ξανά είμαστε στα ίδια όσον αφορά τα, το θέμα αυτό τις διάφορες πτυχές περιβαλλοντικές, κοινωνικές και διαχείρισης. Ο Μάρη, ίσως η, η, θα το έχει στην έκθεσή της. Το αναφέρατε ως λεπτομέρεια. Για μένα δεν είναι λεπτομέρεια. Τι γίνεται με την νομοθεσία ΠΡΕΠΣ. Σε αυτή την νομοθεσία το Κοινοβούλιο, όπως και στο STS και σε άλλα θέματα, να έχει κάτι που αναφέρεται στο περιβάλλον, στη σωστή διακυβέρνηση και στα κοινωνικά θέματα. Δεν θέλει να τα εξετάσει αυτά τα θέματα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έγινε αόριστη διαβούλευση με την ΕΖΑ. Η ΕΖΑ δεν έχει ιδέα για αυτά τα θέματα είπαν δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ήδη αυτό προβλέπεται από την νομοθεσία. Και όταν θα αναφερθείτε στην ιεράρχησή σας και όλα αυτά θα πούν, κοιτάξτε, είναι πέρα από την ε, νομική βάση του ΠΕΠΣ. Και λείπει και χρόνος. Χρειάζεται πολύς χρόνος όλα αυτά να ολοκληρωθούν. Υπάρχει δυναμική, αλλά χρειάζεται και χρόνος. Εδώ μεταξύ έχουμε μια νομική βάση που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, αλλά δεν μπορούμε γιατί περιμένουμε. Παρακαλώ να μας βοηθήσετε να κινηθούμε τώρα, να ξέρουμε ποια είναι η νομική βάση. Τι, αυτό που συμπεριλαμβάνεται στο άρθρο 8.4 της νομοθεσίας ΠΡΕΠ. Φαίνεται λεπτομέρεια, αλλά είναι θέμα νομικής βάσεως που υπάρχει, αλλά δεν τη χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήταν εδώ και ο Παπαδημούλης, αλλά έφυγε. you Ο κύριος Κόμπορν. Μα δεν θα είχα ποτέ την ευκαιρία να μιλήσω. Οι ιδέε τη Ένωση για ένα βιώσιμο χρηματοπιστωτικό σύστημα θα έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα. Οι Ηνωμένε Πολιτείες δεν ενδιαφέρονται. Σε αυτές τις ε, αντιεμπορικές ιδέες σας για αυτό το σύστημα. Γιατί δεν ε, προσανατολίζονται στις ανάγκες της αγοράς ε, και των συναλλαγών. Εμείς ως Βρετανία και οι Αμερικανοί έχουν τέτοια προσέγγιση, όμως δεν είστε. Και αυτό δεν βοηθάει στη δουλειά και όλες αυτές οι ανοησίες για πράσινα ομόλογα. Σήμερα σε κάποιες εφημερίδες αναφέρεται ότι η Βρετανία μπορεί να υπονομεύσει το κοινωνικό πρότυπο της Ευρώπης. Και λέγεται ότι αναέτος μπορεί να κερδίσει 4,7 δίση η Βρετανική οικονομία γιατί δεν θα σέβεται τα όρια εκπομπών. Το έχω συζητήσει με ανθρώπους από το City. Για να υπάρχει σταθερό και βιώσιμο χρηματοπιστωτικό σύστημα χρειάζεται ανταγωνισμός. Αλλιώ δεν υπάρχει βιωσιμότητα. Ενώ το δικό σα σύστημα είναι εντελώ προστατευτικό. Εφόσον εξαιρείτε το, την αγορά χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου, οι κύριοι Μπαρνιέ και Φερχόφστατ, όσο και δεν του αρέσει, θα πρέπει να καταλάβουν ότι το σύνδεσμο του Λονδίνου είναι η χρηματοπιστωτική καρδιά της Ευρώπης. Είμαστε οι τραπεζίτες της Ευρώπης και θα συνεχίσουμε και μετά την αποχώρησή μας. Οι λαοί της Ευρώπης και του Ηνωμένου Βασιλείου θέλουν πραγματικές δουλειές, όχι υποθετικές δουλειές. Και οι πραγματικές δουλειές φασίζονται στην ε, πραγματική οικονομία. Δεν είναι βιώσιμα αυτά τα πράγματα. Είστε σε άλλο πλανήτη. Δεν είστε στον ίδιο πλανήτη με την Κίνα και την Άπα Ανατολή και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν, και η Βρετανία. Δεν είστε στον ίδιο πλανήτη. Ζείτε σε ένα κόσμο της φαντασίας σας. Στην ουσία θα διαλύσετε το χρηματοπιστωτικό τομέα της Ευρώπης. Θα καταρρεύσει γύρω σας. Θα υπάρξει ανεργία, κοινωνική αναταραχή και πολιτική διάλυση. Εμείς φεύγουμε και δεν μας ενδιαφέρουν όλα αυτά. Δεν θέλουμε τέτοιες χρηματοπιστωτικές παλαβομάρες. Γι' αυτό θέλουμε και εσείς να είστε σε καλή κατάσταση για να μπορείτε να αγοράσετε τα προϊόντα μας. Και θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι θα συμπεριληφθούν οι δικές μας χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ε, στο σύστημά σας. Εάν δεν υπάρξει κάτι τέτοιο, κάποιες Ιταλικές τράπεζες μπορεί να φαλυρίσουν. Δεν βοηθάνε όλα αυτά κανέναν. Πρέπει να πείσετε τους κυρίους Φερχόφστατ και Μπαρνιέ να καταλάβουν ότι οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες της Βρετανίας είναι ουσιώδεις για την Ευρώπη. Λοιπόν, άλλος κανείς θέλει το λόγο. Ο Πέτα Ζήμαν. Τώρα είναι δύσκολο να μη σχολιάσω τις βλακίες που μόλις ακούσαμε. Να πω μόνο ένα πράγμα. Οι Βρετανοί και το σύνδετο του Λονδίνου είναι σημαντικά για μένα. Αλλά δεν είναι τόσο σημαντικά ούτως ώστε να καταστρέψουμε τη δική μας οικονομία. Και ναι, θα υπερβούμε, θα καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα για την καταστροφή που προκαλέσατε και θα πληρώσουμε όλοι. Αλλά να μην θεωρείτε ότι είστε σε θέση να μας εκβιάσετε. Και όλες σας οι ομιλίες είναι, ακούγονται ως εκβιαστικές. Αλλά κοιτάξτε, όσο περισσότερο μας προκαλείτε έτσι, τόσο περισσότερο ενισχύεται την ενότητά μας. Αυτά απλώς εισαγωγικά. Ένα σχόλιο τώρα. Αναφερθήκατε στις υποδομές και εγώ νομίζω ότι είναι σωστό να υπάρξει σωστή χρηματοδότηση των υποδομών και μέσω ιδιωτικών επενδύσεων. Αλλά κάτι που διαπίστωσα εξετάζοντας κάποια κείμενα όταν θέλουμε να ευνοήσουμε τη χρηματοδότηση των υποδομών και να μειώσουμε το κόστος της υπάρχει μια προκατάληψη ήδη αρχική υπέρ του ιδιωτικού τομέα. Αλλά εγώ είμαι Γερμανός Στη Γερμανία έχουμε μια μακρά και σωστή παράδοση χρηματοδότηση των υποδομών με δημόσιο χρήμα. Πρέπει λοιπόν να μην υπάρχει για πολιτικούς λόγους προαπόφαση υπέρ των ιδιωτικοποίησεων και να θεωρούμε ότι η ιδιωτική χρηματοδότηση είναι πάντα ευθυνότερη. Πάντα αν υπάρχει ιδιωτική αναχρηματοδότηση είναι πάντα φθηνότερη η χρηματοδότηση των υποδομών. Όχι, στη χώρα μου Είμαστε ιδιαίτερα πεπισμένοι ότι οι δημόσιες υπηρεσίες και οι υποδομές είναι βάση του δημόσιου βίου. Είναι κάτι που θα πρέπει να χρηματοδοτείται από το δημόσιο τομέα και είναι δυνατόν να υπάρξει καλή χρηματοδότηση δημόσια. Δεν είναι κατά ανάγκη καλύτερα να υπάρχει ιδιωτική χρηματοδότηση. Ευχαριστώ πολύ. Η Νίνα Γκίου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ να αποστασιοποιηθώ από τα σχόλια του κ. Κόμπερν. Να επαναλάβω ότι δεν θέση του Ηνωμένου Βασιλείου, της Βρετανίας ή του ΣΥΤΙ. Ευτυχώς στη Βουλή των Κοινοτήτων δεν έχουμε μέλη του UKIP. Και αυτή δεν είναι θέση του Κοινοβουλίου του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Ηνωμένο Βασίλειο θέλει να κινηθεί προς πιο βιώσιμο χρηματοστατικό τομέα και εκτιμά την έκθεση που εκπονήσατε. Οι ερωτήσεις μου δεν σχετίζονται με αυτά. Ερώτηση. Πώς θα έχουμε σαφέστερη εικόνα περί πρασίνου και βιωσιμού. Φαίνεται να υπάρχουν διαφοροποίησεις όσον αφορά το τι περιγράφεται ως πράσινο. Θέλουμε γενικότερη κατανόηση σε παγκόσμιο επίπεδο. Υγείται σε πολλούς από αυτούς τομείς η Κίνα. Πώς μπορούμε να έχουμε σαφέστερη εικόνα και να γνωρίζουμε αν αυτό που κάνουν εκείνοι πραγματικά αφορά τον πράσινο τομέα. Επόμενο σημείο. Η αποκάλυψη των κινδύνων, γνωστοποίηση κινδύνων των σχετιζομένων με το κλίμα. Υπάρχουν κρίσιμες πληροφορίες που χρειάζονται οι επενδυτές Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω τι γίνεται με τις, τα μη χρησιμοποιημένα στοιχεία ενεργητικού που ίσως να ενεργοποιηθούν αύριο τα μη ενεργοποιημένα σήμερα. Πώς μπορούμε να προβλέψουμε την εξέλιξη εκεί. Πώς μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα τι, τι σημαίνει αυτή η έννοια stranded assets. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Ευχαριστώ για τα συγχαρητήρια και τα κομπλιμέντα. Θα τα διαβιβάσω στην ομάδα. Ήταν πράγματι υπέροχη ομάδα και όπως είπες Περβάνς ανταποκρίθηκαν στην πρόκληση και εξέτασαν τα θέματα που σε ενδιαφέρουν. Ακολουθήσω αντίστροφη σειρά απαντήσει. Όσον αφορά την ιεράρχηση των θεμάτων, μια καλή αφετηρία είναι από την υπηρεσία περιβάλλοντος. Είπαν ότι τρία συστήματα δεν λειτουργούν σωστά όσον αφορά θέματα βιωσιμότητας ή κλίματο. Το ενεργειακό σύστημα, το μεταφορικό σύστημα και το σύστημα διατροφής. Το ενεργειακό σύστημα δεν έχει ευθυγραμμιστεί με τη βιωσιμότητα για τους λόγους που ξέρουμε. Γι' αυτό θα είναι εύκολο να εφαρμόσουμε την ιεράρχηση. Υπάρχουν κάποια στοιχεία για τις εκπομπές, το ενεργειακό μείγμα, υπάρχουν νέες τεχνολογίες και το θέμα είναι όλα αυτά πώς θα τα συγκεράσουμε. Όσον αφορά τις μεταφορές και το μεταφορικό σύστημα, γίνονται εκτενείς συζητήσει και θα είναι ευκολότερο να δούμε πού απαιτούνται επενδύσει Σε πολλές χώρες και σε πολλές πόλεις διεξάγεται αυτή η συζήτηση. Το τρίτο σύστημα, το δυσχερέστερο, το, το σύστημα των τροφίμων. Πώς παράγουμε τα τρόφιμα, πώς μεταφέρουμε τα τρόφιμα είναι κάτι που είναι ε, επιβλαβές για το περιβάλλον λόγω υπερβολικών μεταφορών. Αν σκεφτούμε από πού έρχεται το φαγητό που καταναλώνουμε. Άρα πρέπει να αλλάξουμε το αγροτικό σύστημα, σύστημα καλλιεργιών, το σύστημα παραγωγής και μεταφοράς των τροφίμων. Λοιπόν, αυτή η ιεράρχηση των θεμάτων. Στέγαση αφορά περισσότερο την ενεργεία. 70 δισεκατομμύρια απαιτούνται, τα περισσότερα χρήματα θα διατεθούν για την ενέργεια για καλύτερη μόνωση των κτηρίων. Και αυτό θα ενταχθεί στο σύστημα ιεράρχησης. Θα πρέπει να σκεφτούμε και το θέμα της παγκοσμιοποίησης. Η παγκοσμιοποίηση είναι μια διαδικασία. Δεν μπορεί να τη σταματήσει ή να την αντιστρέψει κανείς. Ίσως όμως πρέπει να γίνουν διαφορετικές προσαρμογές, να υπάρξει ντόπια κατανάλωση και καλλιέργεια και ίσως να ωφεληθούν και κάποιες περιοχές που είναι σε μειονεκτική θέση αντί να έχουμε σε τέτοια τεράστια κλίμακα μεταφορές σε όλο τον πλανήτη. Μετά η ε, αποκάλυψη υποβολή πληροφοριών. Είπατε γιατί δεν πάμε σε υποχρεωτικό χαρακτήρα της ε, διαβιβάσεως στοιχείων. Να σας αναφέρω τρεις λόγους για τους οποίους η ομάδα είπε ότι καλύτερα να περάσουμε μία φάση επιθελοντικής βάσης, να δούμε πώς πάμε και μετά με τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο αυτό μεταφράζεται στην νομοθεσία. Υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα, αλλά υπήρξαν τρία επιχειρήματα που ε, ήταν αντίθετα και οδήγησαν στη λύση που περιέχεται στην έκθεση. Κατά τα τρία επιχείρηματα μέθοδο, νομικό κίνδυνο και χρήση. Τα τρία επιχείρηματα. Όσον αφορά τι μεθόδου, είχα το προνόμιο να, να είμαι αντιπράεδρος της ομάδα Κρούση, της Task Force FSP, συζητήσαμε τις μεθόδου, τις σωστέ, και υπάρχουν εργαλεία αλλά όχι μέθοδοι για την ε, βιωσιμότητα των κινδύνων. Έγινε μία ανάλυση ενδεχομένων, μετά θα πρέπει κανείς να εξετάσει ε, την επιχείρησή του, τα μελλοντικά ενδεχόμενα, αλλά εξετάζοντας το μέλλον χρειάζεσαι μεταβλητές, ε, ε, δείκτες κλπ. Είναι μια μέθοδος που είναι καλή για εσωτερικές συζητήσεις, τροφοδοτεί, αλλά δεν είναι αρκετά ακριβής. Δεν σου δίνει ακριβείς απαντήσεις, σου δίνει φάσματα απαντήσεων. Ε, υπάρχει περιθώριο να εμβαθύνουμε σε αυτές τις μεθόδους που είναι καινοφανείς. το δεύτερο θέμα που είχαμε υπόψη μας ήταν η νομική κίνδυνη. Ε, κάθε αποκάλυψη στοιχείων ε, θέτει μια εταιρεία ενώπιον νομικών κινδύνων. Οπότε, ποια είναι η σκέψη, ας πειραματιστούμε πρώτα πριν εκθέσουμε τις επιχειρήσεις ενδεχόμενους νομικούς κινδύνους. Και τρίτον, η χρήση. Όλοι είμαστε υπέρ του να δώσουμε μακροπρόθεσμες πληροφορίες, πιο μακροπρόθεσμες το θέμα είναι ποιος θα χρησιμοποιεί τις πληροφορίες. Αν μιλήσει στι συγμένες εταιρείε, οι αναλυτές που τις επισκέπτονται είναι αναλυτές που έχουν μοντέλα που εστιάζονται επί ενός, δύο ή τριών ετών και αυτό αναφέρεται στην έκθεση. Σήμερα όταν δείτε τους οικονομικούς αναλυτές που αξιολογούν μια εταιρεία και επενδύουν εστιάζονται σε μια περίοδο ενός έτους, δύο ετών, τριών ετών. 75% ε, είναι τρία χρόνια και λιγότερο. 95% των αναλυτών πέντε χρόνια και λιγότερο. Άρα πολύ δύσκολο να βρούμε ανθρώπους που είναι σε θέση αυτές τις πληροφορίες να τις εισαγάγουν στα μοντέλα τους. Γι' αυτό θεωρήσαμε ότι υπάρχει μια διαδικασία εκμάθησης, όχι μόνο πλευράς εταιριών, να υποβάλουν καλύτερα στοιχεία, να μάθουν μεθόδους, να αισθάνονται ασφαλείς νομικώς, αλλά και για εκείνους που χρησιμοποιούν τις πληροφορίες να επεκτείνουν τα μοντέλα τους. Και αυτό αφορά και τους οίκους αξιολόγησης, τους χρηματοσυντικούς αναλυτές κλπ. Αυτό οδήγησε στο συμβιβασμό, αν θέλετε. Ας χρησιμοποιήσουμε για δύο χρόνια το σύστημα, πειραματιστούν οι εταιρείε και για πολλέ εταιρείε αυτό είναι κάτι καινούριο. Περάσαμε πολύ χρόνο συνομιλώντα με επιχειρήσει στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία πιο συγκεκριμένα. Αυτό ήταν το τομέα στον οποίο εξετέθην. Για πολλού αυτά ήταν καινούργια. Πολλοί είπαν μπορούμε να το εξετάσουμε αυτό, αλλά δεν ξέρουμε. Ποτέ δεν φτιάξαμε ένα σενάριο να δούμε πώ λειτουργεί το σύστημα, ποιο το κάνει, ποιε μεθόδου χρησιμοποιούμε, IWWF κλπ. Άρα είναι μια καμπύλη εκμάθησης που ακολουθείτε. Για το PRIPS καταλαβαίνω αυτό που είπατε, θα το λάβω υπόψη μου στους συζητήσεων της Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί η βαθμολόγηση είπατε ότι με την ΕΣΑ δεν είναι εύκολα τα πράγματα ε, και εμείς ε, ανταλλάξαμε απόψεις με το φορέα. Πιστεύω ότι κατανοούν ότι δεν είναι ουδέτερη αγορά η αγορά δεν λαμβάνει υπόψη επαρκώς τους κινδύνους βιωσιμότητας. Οπότε η βαθμολόγηση βάση των αγορών δεν ευθυγραμμίζεται τέλεια με αυτό που θέλουμε. Και γι' αυτό είναι τόσο σημαντική η δουλειά που κάνουμε. Ε, ίσως δεν θα έπρεπε, δεν μπορώ να αντισταθώ. Όμως στην κατηγορία για τη χρησιμοποιούμε, ζούμε στο φανταστικό κόσμο. Το απορρίπτω. Είχα το προνόμιο να εργαστώ ε, στον εμπορικό τομέα, σε εμπορική επιχείρηση και βιώσιμη επιχειρηματικότητα σημαίνει καλύτερη επιχείρηση. Για τον ασφαλιστικό τομέα αυτό το θέμα τη βιωσιμότητα οδήγησε σε πολύ αυστηρό προβληματισμό περί καλύτερη προστασίας των εταιριών κατά κινδύνων που απορρέουν το κλίμα, καλύτερων επενδύσεων, καλύτερη κατανόηση των κλιματολογικών κινδύνων, στη μόρφωση μοντέλων κλπ. Πώ μπορούμε να προσανατολίσουμε καλύτερα το ισοζυγείο μα, αν θέλετε, πώς να χρησιμοποιήσουμε μη ενεργοποιημένα στοιχεία ενεργητικού. Το επίπεδο ευαισθητοποίησεως αυξήθηκε και η βιωσιμότητα στην επιχειρηματικότητα ε, λαμβάνεται υπόψη και το επιχειρήν στα πλαίσια βιωσιμότητα είναι καλύτερο επιχειρήν. Όσον αφορά τι υποδομέ, κατανοώ την προσέγγιση σα που έρχομαι από την ίδια χώρα, κατανοώ αυτό που είπατε, το εκτιμώ, αλλά ε, δεν πρέπει να την δούμε σαν ενιαία την υποδομή. Υπάρχουν υποδομές έτοιμε, για ιδιωτικέ επενδύσεις. Ας πούμε, υπεράκτια, σε αιωλικές εγκαταστάσεις. Για κάποια κράτη-μέλη έχουν προχωρήσει, το εφαρμόζουν αυτό, άλλες χώρες όχι. Είναι πολύ δύσκολο να επενδύσουν στις νέες τεχνολογίες. Αν μιλήσετε την, ε, με κάποια πόλη που είναι μακριά, βόρεια, νότια, ανατολικά στην Ευρώπη, θα θέλαν να μάθουν την εμπειρία για ε, ε υπεράκτιες αιωλικές εγκαταστάσεις. δεν υπάρχει κάποιος στην Ευρώπη που μπορεί να δώσει, να μεταδιδάσει την ε, τεχνογνωσία. Να ξέρουμε στη Γερμανία αυτό λειτουργεί, αυτό λειτουργεί, στη Γαλλία αυτό λειτουργεί, αυτό λειτουργεί. Μπορείτε σε αυτή την απόσταση να βάλετε αιωλική μονάδα, τάδε μεγέθου κλπ. Λείπει ε, η συμβουλή τεχνική, μη εμπορική φύσεω. Ένα μικρό φορέα ε, σε αυτό το τομέα θα ήταν κρισιμότατος να βοηθήσει τα κράτη-μέλη να προσαρμοστούν και να μάθουν από τις εμπειρίε άλλων χωρών τη Ευρώπη. Δεν μπορούμε να κρίνουμε αν χρειάζεται ιδιωτικό ή ε, δημόσιο τομέα. Στον ιδιωτικό τομέα είναι το θέμα πώ μπορούμε να βοηθήσουμε τι επιχειρήσει να συντονιστούν με τα τεκτενόμενα στην τεχνολογία. Ε, ακροθυγός κάποια τελευταία σημεία. Κάποια θέματα ιεράρχησα συζήτησα, αποκάλυψη στοιχείων το συζήτησα, επιδοτήσει, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Είναι κάποια θέματα που θεωρούσαμε ότι ήταν εκτό ε, εντολή Ευρωπαϊκή Τάπεζα Επενδύσεων, δανειοδότηση, πολιτική δανειοδότηση. Δεν είμαστε μονάδα αξιολόγηση Ευρωπαϊκή Τάπεζα Επενδύσεων, δεν είμαστε ε, μονάδα αξιολόγηση πολιτική Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτά πρέπει να τα αφήσουμε στην Ευρωπαϊκή Τάπεζα Επενδύσεων, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να τα κάνουν όλα αυτά. Ε, θεωρήσαμε ότι τα θέματα επιδοτήσεων ήταν εκτό τη εντολή μα. Να αναφέρω κανένα δύο σημεία ακόμα. Α, Γεωργία. Ευχαριστώ πολύ, συμφωνώ απολύτω. Η βιώσιμη γεωργία είναι οικονομικά βιώσιμη. Γνωρίζουμε πολλά προγράμματα, έργα που προωθούν βιολογικές καλλιέργειες, βιολογική γεωργία και υπάρχει μεγάλη απόδοση, υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Αυτό το μοντέλο είναι βιώσιμο, τα όλα μοντέλα δεν είναι βιώσιμα. Ναι, από την εμπειρία στη χώρα σας ε, αναφερθήκατε σε σύντομο κύκλο καλλιέργειας απόδοσης. Αυτά και καλό για το περιβάλλον. Για τους χρηματοπιστωτικούς φορολογικούς κανόνες, σωστά, IFRS 2 ε, κλπ. Γενικά, τι, πού πάμε από εδώ και πέρα, τι λαμβάνουμε υπόψη. Ελπίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το οποίο συνεργαστήκαμε στενά ότι θα λάβει υπόψη τι πολλέ από τι συστάσει. Βέβαια δεν μπορούν να συμπεριλάβουν όλε, αυτό είναι σαφέ. Ελπίζουμε ότι πολλά ειδικά συστήματα για λογιστικά, τραπεζικά θέματα τελικά θα συμπεριληφθούν. Δεν θέλουμε να ξανανοίξουμε κεφάλαια, αλλά στην επόμενη ευκαιρία απλώς να αλλάξουμε την προσέγγιση ανάμεσα πω στη βιωσιμότητα, ώστε να έχουμε περισσότερη δανειοδότηση, περισσότερε απασχόλησει και περισσότερη ανάπτυξη στην ευρωπαϊκή οικονομία. Κοινωνικέ υποδομέ. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Α, προσπαθήσαμε λοιπόν να το εξετάσουμε και αυτό που είναι ενδιαφέρον, εξετάσαμε τις κοινωνικές επιχειρήσεις, κοινωνικές υποδομές και υπήρχε ένα θέμα που τονίζουμε η ε, χωρική διάσταση. Ε, η βιώσιμη χρηματοπιστωτική προσέγγιση σημαίνει ναι, ότι ικανοποιούμε το Μιλάνο, το, τη Φραγκφούρτη, το Λουξεμβούργο κλπ. Σημαίνει βιώσιμο χρηματοστικό, ε, χρηματοστικό τομέα να δώσουμε κεφάλαιο στι περιφέρειε του Βορρά, του Νότου, τη Ανατολή, τη Δύση, όπου ο κόσμο φεύγει από εκεί. Αν δείτε τι πληθυσμιακέ μετακινήσει στη Λιθουανία, Φερρυπίν, Ανατολική Γερμανία, Νότια Ιταλία, Ισπανία. Ε, θα ήταν πολύ σημαντικό ο βιώσιμος χρηματοστικός τομέας να καταφέρει να δώσει κεφάλαιο κυρίως σε κοινωνικές υποδομές σε περιοχές που είναι απομακρυσμένες περιοχές όπως αποκαλούνται. Οπότε δεν είναι για περισσότερο εμπόριο ε, στο χρηματιστήριο, αλλά να προωθηθεί βιώσιμη διάσταση, να δώσουμε επενδύσει θέσει απασχόληση σε απομακρυσμένε περιοχέ, να βοηθήσουμε τι ε, περιοχέ να αναπτυχθούν. Αυτή αυτή είναι η χωρική διάσταση ε, του ε, βιωσίμου χρηματοστοτικού τομέα. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι ολοκληρώσαμε τις εργασίες μας, πέρασε η ώρα. Θέλετε να πείτε κάτι. Κοιτάξτε, έπρεπε να τελειώσουμε στις 11. Είναι 11 και 5. Πλούσια. Χρήσιμη συζήτηση. Συγχαρητήρια για το έργο σας. Και έχουμε και άλλες πληροφορίες, η ζωή πληροφοριών για την έκθεσή μας. Ελπίζουμε να συμβάλλουμε και εμείς και να εντάξουμε διάφορα στοιχεία με κάποιο τρόπο στην ομοθεσία. Διάβασα με ικανοποίηση, με χαρά την παράγραφό σας στη σελίδα 68 για μείωση κεφαλοχικών απαιτήσεων για δανειοδότηση του πράσινου τομέα. Αυτό κάναμε στην έκθεση σήμερα. Αισθανόμαστε δικαιωμένοι στην αποφασιστικότητα που δείξαμε. Αλλά δεν υπάρχει ένα και μοναδικό μέτρο που λειτουργήσει από μόνο του. Μιλάμε για συνδυασμό μέτρων. Θέλουμε στοχευμένα μέτρα. Θέλουμε σφαιρική εικόνα, διάδραση μεταξύ στοιχείων. Αυτό δίνει προστιθέμενη αξία στην έκθεση. Και αυτή είναι η προσέγγιση που πρέπει να ακολουθήσουμε. Με συνέπεια, φιλοδοξία και πρακτικό πνεύμα. Ούτω ώστε να πετύχουμε στόχους που είναι στόχοι μεμονωμένων μέτρων, στα πλαίσια όμως ενός ευρυτέρου πλαισίου και σχεδίου. Ευχαριστώ πολύ. Πέρασε η συνεδριά σας. Γεια σας.